Ε, ότι η Επιτροπή Δεταρρυθμιστών ε, και συντηρητικών έχει προτείνει κάποια ονόματα για να συμμετάσχουν σε αντιπροσωπείς αυτά θα σας ε, δοθούν θα σας διανεμηθούν αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για αυτούς τους διορισμούς θεωρούμε ότι εγκρίνονται οι προτάσεις αυτές τώρα λοιπόν